πυρηνικό τομέα με το ε, Ιράν. Συνεχίζουμε τις επαφές, ε, δεν είναι όμως μυστικό ότι η επιβίωση της συμφωνίας αυτής έχει καταστεί πολύ δύσκολη. Να πω ότι θα υπάρξει μια κοινή επιτροπή με το Ιράν σε επίπεδο ε, διευθυντών στις 6 Δεκεμβρίου σε συνεργασία ή μάλλον ε, προσπαθώ να συντονίσω και τις ε, υπηρεσίες της Επιτροπής που ασχολούνται με το θέμα της πυρηνικής συμφωνίας έτσι ώστε να κρατήσουμε φυσικά και την ενότητα της ευρωπαϊκής πλευράς αλλά και όλων των άλλων συμμετεχόντων στην ε, συμφωνία αυτή. Πιστεύω λοιπόν ότι η ενότητα αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση της συμφωνίας. Συμφωνήσαμε άλλωστε εδώ και λίγες εβδομάδες ότι θα πρέπει να κάνουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε προσπάθεια ε, για να ευοδοθεί η προσπάθεια αυτή και εδώ θέλω να ευχηθώ στον διάδοχό μου ε, κάθε επιτυχία. Και τρίτον, να μιλήσω για το Λίβανο, όπου οι διαμαρτυρίες οδήγησαν στην παρέτηση του Πρωθυπουργού. Ο Λίβανος είναι ένα ειδικό εταίρος και έχει μια ειδική θέση στην καρδιά μας. Ο κόσμος στον Λίβανο ζητάει σωστή και δίκαιη διακυβέρνηση και είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας εμπνεύσει γιατί δείχνει πόσο ανοιχτή είναι η κοινωνία του Λιβάνου. Πρέπει να διατηρηθεί η ειρήνη και η σταθερότητα η οποία χαρακτηρίζει τη χώρα αυτή όλα αυτά τα χρόνια. Πρέπει να υπάρξει ταχύτατα μία λειτουργική κυβέρνηση, πρέπει να υπάρξει μία αποφασιστική και γρήγορη εφαρμογή των μέτρων κατά της διαφθοράς σύμφωνα με τις προσδοκίες του λαού του Λιβάνου είναι μια ευκαιρία έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχει ανάγκη η χώρα διατηρώντας τη σταθερότητα όμως ταυτόχρονα της χώρας αυτής. Κάτι άλλο τώρα που δεν άπτεται άμεσα το η σημερινή συζήτηση, να μην ξεχνάμε ότι το σύνολο της Μέσης Ανατολής είναι μια πάρα πολύ ευαίσθητη περιοχή. Παλαιστίνη δεν ξεχνάμε την κατάσταση στη Συρία, δεν έχει ρυθμιστεί ακόμα, το αντίθετο στην βορειοδυτική η κατάσταση έχει χειροτερεύσει δυστυχώς ε, μετά ε, λίγες εβδομάδες ε, την ε, εισβολή των Τούρκων τις, μετά λίγες εβδομάδες από την εισβολή των Τούρκων στην νοτιοανατολική Συρία. Γίνονται προσπάθειες έτσι ώστε να ηρεμήσει κάπως η κατάσταση και να βελτιωθούν οι δύο διεπικοινωνίες. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε πολυμερείς τρόπους συνεννόησης Συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας όπως το Ιράκ, ο Λίβανος, να σταθεροποιήσουμε ακόμα περισσότερο τις χώρες αυτές και να τις βοηθήσουμε οικονομικά. Κάθε μία από αυτές τις χώρες θα πρέπει να βρει τον δικό της δρόμο, όμως κανένας δεν μπορεί να τους το δώσει αυτό, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει τον διάλογο και την συνοδεία των μέτρων αυτών. Είναι μια περιοχή για την οποία ε, φροντίζουμε ιδιαίτερα και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ένας αξιόπιστος εταίρος, ένας εταίρος ειρήνης. Ευχαριστούμε κύριε Μουγκερίνη. Εκ μέρους ε, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Στέφανετς, τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τις τελευταίες διαδηλώσεις ε, και διαμάχες στο Ιράν. Αυτές οι διαμαρτυρίες ε, εδώ και 11 μέρες και στις 31 επαρχίες του Ιράν σε πάνω από 176 πόλεις ε, όπως ανακοίνωσε η αντιπολίτευση από 400, οδήγησαν σε πάνω από 450 νεκρούς αλλά μπορεί να είναι και περισσότεροι αυτοί που δολοφονήθηκαν ε, με βία από τις Ιρανικές ε, δυνάμεις ασφαλείας. Είναι θλιβερός ο κατάλογος. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται ο 14χρονος Νίκτας Φαντάνη. Στην ε, περίπτωση αυτή, αυτού του κοριτσιού της είπαν οι αρχές ότι επειδή ήταν μόλις 14 ετών δεν θα καλύψουν το κόστος της κηδείας. Είναι απίστευτο η κυβέρνηση του Πρόεδρου Ροχάνη που θεωρείται μετριοπαθής έκλεισε το ίντερνετ για να απαγορεύσει να κυκλοφορήσουν ειδήσει και βίντεο από αυτά τα εγκλήματα και να βγουν από το Ιράν. Η κυβέρνηση επίσης αρνείται να δώσει τα ε, σώματα στις οικογένειες και απαγορεύει τις κοιτίες. Ανησυχώ για το τι θα γίνει ε, με τους κρατούμενους και πώς θα τι μεταχείριση θα την χάνουν. Κάποιοι αξιωματούχοι είπαν ότι πολλοί από αυτού που έχουν συλληφθεί θα εκτελεστούν σύντομα με ε, δημόσιο απαγχωνισμό. Ε, ειδικότερα τα μέλη της PMOI, ε, της αντιστασιακής οργάνωσης που κατηγορεί η κυβέρνηση για την ανταρσία. Τα εγκλήματα της Ιρανικής κυβέρνησης είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αναμφίβολα. Ε, εναντίον ανθρώπων που υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους ε, στον δρόμο και δεν υπάρχει ε, δεν έχει δικαίωμα η κυβέρνηση να τους λαμβάνει και να τους σκοτώνει. Η κυρία Ρατζάβη, αρχηγός της αντιπολίτευσης, απευθύνει έκκληση προ τα Ηνωμένα Έθνη να αποστείλει ανθρωπιστικέ αποστολέ των παρατηρητών στο Ιράν για να διαπιστώσουν τα εγκλήματα που διαπράττει η Ιρανική κυβέρνηση. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του Ιρανικού λαού και παροτρύνω την είπατε εκπρόσωπο να πράξει το ίδιο να σταματήσει η σημερινή πολιτική διότι κατά την απόψή μου αυτή έχει αποτύχει. Δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ζημιώνει την αξιοπιστία της Ευρώπης ε, στα μάτια του Ιρανικού λαού αλλά και στα μάτια ολόκληρου του κόσμου. Οι άνθρωποι μας ε, παρακολουθούν, αναμένουν τη δική μας δράση και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δράσει άμεσα. Ευχαριστώ πολύ. On behalf of Εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών, τώρα η κυρία Σάντος για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπουμε ε, πολιτικά κινήματα. Η κατάσταση στο Ιράν είναι τόσο δύσκολη και τόσο απρόβλεπτη. Δεν μπορούμε να γενικεύουμε και δεν μπορούμε να απλοποιούμε. Μπορούμε να εντοπίσουμε ε, επίπεδα φτώχειας, ε, κακές ε, συνθήκες, διαφθορά, να μην υπάρχει προοπτική για τους νέους. Αυτά είναι τα κοινά σημεία που οδηγούν συνήθως σε εντάσεις. Είτε μιλάμε για το Ιράκ, είτε μιλάμε για το Ιράν, είτε μιλάμε για το Λίβανο. Πρόκειται για χώρες που έχουν εσωτερικά προβλήματα και κρίσεις, οι οποίες βέβαια μεγαλώνουν και ενισχύονται και από εξωτερικούς παράγοντες. Η βία βέβαια σε βάρος των διαδηλατών ε, στο Λίβανο ή αλλού είναι κάτι που καταδικάζουμε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο ούτε στην περίπτωση του Ιράν ε, και την καταστολή που επιβάλλει σε ειρηνικές διαδηλώσεις ή την απαγόρευση του ίντερνετ της ε, αυθαίρετες κρατήσεις και βασανισμούς ή τους ε, θανάτες, τους εκατοντάδες θανάτους. Όλα αυτά είναι απαράδεκτα και ένα πράγμα μπορούμε να πούμε ότι οδηγούν σε ακόμα χειρότερη οικονομική κρίση. Και για το Ιράκ. Εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιδράσουμε και να σταματήσει οποιαδήποτε μεταφορά τεχνολογίας που μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιες βίες καταστάσεις. Ευχαριστούμε εκ μέρους του Ρινιού Γκέτα, ο κύριος Γκέτα για δύο λεπτά. Το αίμα ρέει στη Βαγδάτη, στην Τεχεράνη και αλλού. Τώρα είμαστε μπροστά σε μια νέα Μέση Ανατολή. Ας δούμε καταρχήν στη Βαγδάτη και στη Βηρητό τις διαδηλώσεις. Εκεί δεν υπάρχουν ε, Κούρδοι, Σίτες, Σουνίτες κτλ. Υπάρχουν εδώ Λιβανέζοι, εδώ Ιρακινοί, ε, πολίτες των χωρών αυτών που χέρι-χέρι διαμαρτύρονται για την επιδείνωση των συνθηκών ζωή τους, για το εύρος της διαφθοράς και κανείς ε, δεν θα το έλεγε ότι τα σύνορα ανάμεσα στις διαφορές κοινότητες που συνυπάρχουν θα καταργούνταν τόσο εύκολα σε αυτές τις χώρες. Πρόκειται για χώρες που γίνονται έθνη. Και τις τελευταίες εβδομάδες φάνηκε ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες και το Ιράν. Ε, στο Λίβανο αμφισβητείται και Εσβολά όπως ε, και τα άλλα κόμματα και στο Ιράκ όλες οι συνδικές οργανώσεις καταδικάζουν το κράτος. Πρόκειται για δύο χώρες που διαμαρτύρονται για το προτεκτοράτο που θέλει να τους υποβάλει το να τους επιβάλλει το Ιράν. Και είναι πολύ σοβαρό όταν οι ίδιοι οι Ιρανοί διαμαρτύρονται για την αύξηση των τιμών και για την ενίσχυση της τοκρατίας. Εδώ και 20 χρόνια λοιπόν ε, πάει από τη μία κρίση στην άλλη το καθεστώς εκεί, αλλά με ρυθμό που επιταχύνεται και το βάθος διευρύνεται. Έτσι λοιπόν η κατάσταση αυτή στη Μέση Ανατολή δεν είναι όπως ήταν και όλα θα μπορούσαν να αλλάξουν στην περιοχή αυτή όπου τροποποιούνται οι ισορροπίες κάθε μήνα. Και όλα αυτά συμβαίνουν δίπλα μας αγαπητοί συνάδελφοι. Περισσότερο από ποτέ θα έπρεπε κανείς να είναι κούφος και τυφλός για να μην βλέπει ότι η Ένωσή μας πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα μιας υπερδύναμης για να έχει λόγο στην περιοχή. Ευχαριστούμε κύριε Γκέτα. Επόμενος ομιλητής, η κύριε Νόημαν, εκ μέρους των Πρασίνων της Ελευθερής Συμμαχίας. Για τρία λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν 30 χρόνια οι άνθρωποι κατέβαιναν στους δρόμους στην Ευρώπη για να υπερασπίσουν την ελευθερία και τη δημοκρατία δεν ήταν οργανωμένοι, αλλά ήταν ενωμένοι σε μία απέτηση. Εμείς είμαστε ο λαός και πριν δύο εβδομάδες εδώ συγχαρήκατε τους εαυτούς σας για τις επιτυχείς ε, διαδηλώσεις και πώς άλλαξαν αυτά τις ζωές μας προς το καλύτερο. Από φέτος το καλοκαίρι έχουμε διαδηλώσει σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, στην Αλγερία. Συνεχίζονται στην Αίγυπτο βίαιη καταστολή στο Λίβανο, παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργό ε, στο Ιράκ, διαμαρτυρίες ε, που έτυχαν τεράστιας βίας, 350 ε, έχασαν τη ζωή τους, Ιράκ, τεράστιο blackout των μέσων, δεν έχουμε καν αξιόπιστες πληροφορίες, αλλά πάνω από 100 έχουν χάσει τη ζωή τους, είναι βέβαιο. Σε όλες αυτές τις εξεγέρσεις βλέπουμε ανθρώπους να κατεβαίνουν στους δρόμους για να ε, υπερασπιστούν τις αξιώσεις τους ε, κατά της ε, διαφθοράς, της καταστολής, υπέρ της δημοκρατίας και τι νέο υπάρχει σε αυτές τις διαμαρτυρίες ότι δεν τους ενδιαφέρει πλέον σε τα όρια μεταξύ λαών ή ιδεολογιών. Λένε είμαστε όλοι Ιρακινοί. Αυτό φωνάζουν στους δρόμους της Βαγδάτης και αυτό τρομάζει. Ε, μια 17χρονη ε, έχασε τη ζωή της με δακρυγόνα στη Βαγδάτη, μια μητέρα ε, στο Κάιρο ε, διαμαρτύρει, διαδηλωτές με λουλούδια και τους έριξαν ζωντανά πειρά στο Ιράν και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις έχουμε γιορτάσει 30 χρόνια ειρηνικής επανάστασης και παρακολουθούμε άπραγοι για άλλη μια φορά στο Ιράκ. Είχαμε παρουσίαση για χρόνια, του έχουμε υποστηρίξει με ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουμε έργα νοικοδόμηση. Έχουμε μία αποστολή για την ασφάλεια, για τη μεταρρύθμιση του τομέα τη ασφάλεια στην ίδια χώρα αυτή όπου δεν υπάρχουν γιατροί για του ε, τραυματίε, όπου ε, πυροβολούν ειρηνικού διαδηλωτέ και στου δρόμου του Ιράκ αρνούνται την παρέμβαση του Ιράν οι ΙΠΑ έχουν χάσει την αξιοπιστία τους και διαμάρτη και οι διαδηλωτέ απευθύνουν έκκληση προς εμάς, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύψουμε το κενό που άφησαν οι ΙΠΑ, να οργανώσουμε διάλογο, να σταματήσουμε τις δολοφονίες, να ερευνήσουμε τις καταχρήσεις, να γίνει μια πραγματική μεταρρυθμίση του τομέα της ασφάλειας και να τους μάθουμε τη χρηστή διακυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση εκδίδει διάφορες δηλώσεις χωρίς καμία δέσμευση. Ας είμαι σαφής, συναδέλφοι. Το να κάνουμε τίποτα, το να μένουμε άπραγοι, δεν κάνει παρά να επιδεινώνει τις καταστάσεις αυτές. Έχουμε προδώσει ήδη τους διαδηλωτές της Αραβικής Άνοιξης το 2011. Δεν πρέπει να τους προδώσουμε ξανά. Είμαστε όλοι άνθρωποι με ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Thank you. On behalf of the... Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ριβιέρ από την Ταυτότητα και Δημοκρατία. Υπάρχουν συνεχείς εξωτερικές παρεμβάσεις και περιφερειακές επεμβάσεις στη χώρα. Η σταθεροποίηση μετά από την Αμερικανική παρέμβαση δεν εμποδίζει το Ιράκ να συνεχίσει να διαλύεται που είχε πνιγεί από ένα ολοκληρωτικό καθεστώς αλλά δυστυχώς και μετά την Αμερικανική παρέμβαση υπήρξε η καταστολή της επιθυμίας του λαού να ε, βρει ε, την ελευθερία του και οι ανόητες παρεμβάσεις μας ε, οδηγούν στο χάος. Ο Μοντεσκιό έλεγε ότι θα πρέπει να ακουμπάμε τους νόμους μόνο με τρεμάμενο χέρι. Ας βοηθήσουμε το Λίβανο από την περιοχή αυτή της Μέσης Ανατολής που μας έδωσε τον μονοθεϊσμό αλλά και τη γεωργία. Οι κάτοικοι του Λιβάνου έχουν διεκδικήσει αυστηρά δικές τους. Βλέπουμε ότι υπάρχουν μόνο σημαίες του Λιβάνου στις διαδηλώσεις αυτές. Είναι μήνυμα ελπίδας. Ας μην χειροτερεύσουμε την κατάσταση και να πρέπει να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή να συνεχίσει με το καθεστώς ισορροπίας των διαφορετικών ομολογιών. Ο Λίβανος είναι η καλύτερη απάντηση στην φαρβαρότητα του Ντάεσ. Τώρα θα πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν τον κόσμο που έχει ανάγκη και να υπερασπιστούμε τον πλουραλισμό. εξ ονόματος των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών η κυρία Φώτιγκα. Ευχαριστώ. Υπάρχουν ίχνοι των παρεμβάσεων του Ιράν σε όλη την περιοχή, σε κάθε σύγκρουση, σε κάθε πόλεμο και η παρουσία αυτή φυσικά είναι εις βάρος της σταθερότητας και της ειρήνης αλλά οι χειρότερες παρεμβάσεις φυσικά ελήφθησαν εις βάρος της πολυεθνοτικής και ποικίλη ε, σύνθεσης ε, του λαού του Ιράν τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση των Μολάδων ε, εδώ και δύο χρόνια εις βάρος των διαμαρτυρωμένων μαζικές οι διαμαρτυρίες και στις 31 επαρχίες και στην πλειοψηφία των μεγάλων πόλεων. Διεκόπη η λειτουργία του ίντερνετ και συνεχίζονται ε, γεμάτη βαρβαρότητα, γεμάτες βαρβαρότητα επιθέσεις εναντίον του πληθυσμού. Έχουν υπάρξει ήδη 300 νεκροί τις τελευταίες 11 μέρες και πάνω από 10.000 συλλήψεις και θα πρέπει να ανησυχήσουμε για την κατάστασή τους. όπως ακριβώς είχε συμβεί και παλαιότερα με τους πολιτικούς κρατουμένους. Η μοίρα τους ε, είναι ακριβώς καρπός των εγκλημάτων των δικαστικού σώματος στο Ιράν. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν από το διεθνές δίκαιο να σταματήσουμε να χαμογελάμε στους μολάδες και να αντιδράσουμε. Εξ ονόματος της ενιαίας Ευρωπαϊκής και Πράσινης Αριστεράς η κυρία Έρνστε 1,5 λεπτό. Αυτό που βλέπουμε στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες εβδομάδες είναι τραγωδία. Το ότι στο Ιράν χιλιάδες κατέβηκαν με κοινωνικές απαιτήσει ε, στους δρόμους ε, ήταν δικαίωμά τους. Παρά τις απαγορεύσεις διαδηλώσεων, παρά ε, της καταπολέμησης των ελευθεριών με μεγάλο θάρρος και κόστισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους δεν μπορείς να πυροβολείς διαδηλωτές, πρέπει να το πούμε καθαρά, ο θάνατος ανθρώπων δεν μπορεί να είναι μια παραπλευρή ζημία, όποιος και αν είναι ο λόγος. Και έτσι λοιπόν εγώ εδώ αρνούμε, εξ ονόματος της ομάδας μου, αρνούμε ε, να ξεχάσω τους διαδηλωτές, ε, τους άνδρες, τις γυναίκες, ε, τους γονείς, τα παιδιά και κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της ε, αντιπροσωπής για το Ιράν που προεδρεύω θέλω να σας παροτρύνω να γράψετε ε, μια επιστολή στους συναδέλφους σας, ομολόγους σας στο Ιράν, στο Ιρανικό Κοινοβούλιο γιατί με τις απόψεις ότι όχι μόνο πρέπει να αντιδράσει η Κομισιόν αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό αναμένεται από εσάς. Είναι ντροπή εμείς ως Ευρωπαίοι να μην κάνουμε κάτι αποτελεσματικό για να σταματήσουν οι τρομακτικές κυρώσεις στον ΗΠΑ. Προφανώς ε, μας είναι πολύτιμες οι διατλαντικές σχέσεις, αλλά δεν μπορούμε να πουλάμε το μέλλον του Ιράν. Είναι σημαντικό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και δεν πρέπει, πρέπει να έχουμε μια θαραλέα ευρωπαϊκή πολιτική και να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Ευχαριστούμε από τα ανεξάρτητα μέλη, από τους μη εγγεγραμμένους, ο κύριος Καστάλντο, 1,5 λεπτό. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω στα μέλη ότι πρέπει να τηρούν το χρόνο αγόρευση και με βέβαια θα το κάνετε γιατί είστε και αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ συνάδελφε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι τόσο περίπλοκη που χρειάζεται να την εξετάσουμε πιο δομημένα. Αφενό υπάρχει μια κρίση διάχυτη ε, στη Μέση Ανατολή. Αλλά οι ιδιαιτερότητε κάθε χώρα απαιτούν ε, συγκεκριμένε επιμέρου συζητήσει. Θα επικεντρωθώ σε μια χώρα που με αφορά ιδιαίτερα ε, σημαντική στρατηγικά ε, για την περιοχή στο Λίβανο. Η βεριτόσα αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου κρίση πολιτική και οικονομική με χρέος 150% του ΑΕΠ, πληθωρισμό εκτός ελέγχου και εισοδήματα πάρα πολύ χαμηλά και μια οικονομία στο πλαίσιο της κατάρρευσης. Ε, στα πρόθερα της κατάρρευσης, ε, αδύνατες μεταρρυθμίσεις λόγω της πολύπλοκης ε, πολιτικής κατάστασης, ειδικά μετά από την παρέτηση του Πρωθυπουργού Χαρίρη και τη δυσκολία σχηματισμού νέας κυβέρνησης. Αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζουμε όλοι πόσο είναι κρίσιμη σημασία γεωπολιτικά αυτή η χώρα και πόσο τεράστιε θα είναι οι συνέπειε σε περίπτωση σταθεροποίηση του. Μία νέα κυβέρνηση θα πρέπει να δεσμευτεί για τι απαραίτητε οικονομικέ μεταρρυθμίσει και να καταπολεμήσει τη διαφθορά που παραμένει μία από τις αιτίες που οδήγησε στις σημερινές διαδηλώσεις. Αλλά ο Λίβανος δεν θα βγει ποτέ από αυτή την κρίση αν συνεχιστεί αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Σήμερα υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες στο Λίβανο. Χρειάζεται ε, μεγαλύτερη, σημαντικότερη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτή που παρέχουμε μέχρι τώρα. Οπότε καλώ την Νέα Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα ως κατεπήγον. Ε, αν δεν παρεύουμε θα υπάρξουν απρόβλεπτες και σίγουρα δραματικές συνέπειες. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Κιμπουρόπουλος, παρακαλώ. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι σε αυτή την αίθουσα έχουμε υπάρξει υπερβολική για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς η ευρώπη οφείλει να είναι ο φάρος δημοκρατίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ανάπτυξης διεθνώς. Όμως είναι αλήθεια ότι είμαστε ιδεαλιστές. Θα θέλαμε πολύ η ευρύτερη Μέση Ανατολή, η γειτονιά μας, να μοιράζεται τις ίδιες αξίες με εμά απέναντι στις γυναίκες, τα παιδιά, τους νέους, τους ανάπηρους, αλλά και τους αντιφρονούντες, τους αλόπιστους και τις διαφορετικές εθνότητες. Όμως άλλο Σουηδία και Ελλάδα και άλλο Αίγυπτος και Συρία. Από τον ενθουσιασμό μας, κάποτε μπορεί να υποστηρίξαμε και κάποιες ζωηρές επαναστάσεις που έφεραν πολύ, πολύ χειρότερα καθεστώτα από τα αρχικώς αναπτραπέτα. Άρα, έχουμε πλέον μάθει πως ο ιδεαλισμός πρέπει να εξισορροπείται με λίγο ρεαλισμό και εικόνα του αποτελέσματος. Πρέπει να πονηρευτούμε, καθώς παράγοντες αστάθειας δούνε στην ευρύτερη Μέση Ανατολή παραμονεύοντας να εγκαταστήσουν σκληρά οπισθοδρομικά καθεστώτα. Με όσες δυναμίες και αν έχουν, η Αίγυπτος και το Ισραήλ είναι βράχοι φιλίας και πλέον σταθερή και αξιόπιστοι εταίροι της Ευρώπης στη Μέση Ανατολή. Και γνωρίζουμε καλά ότι οι αφότεροι φέρουν την πρόθεση της αυτοβελτίωσης. Αναφορικά με το Ιράκ, φοβάμαι ότι όσο δεν στηρίζουμε δυναμικά την ανοικοδόμησή του, θα το μετανιώνουμε. 11 από τα 36 εκατομμύρια της χώρας χρήζουν άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δυνητικοί πρόσφυγες. Μπορεί να μην βρίσκονται ακόμα στην ευρωπαϊκή γη, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο καθένας από εσάς μπορεί να καταλάβει το πατέρα και τη μητέρα που θα κάνει τα πάντα για να σώσει το παιδί του. Και αυτοί θα αποτελέσουν την κύρια μάζα του ξεριζωμού. Είμαι σίγουρος ότι πέραν τη ανάσχεση της προσφυγιάς, ο αθλητισμό μας κινεί να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Πολλούς παραξενεύει ο μεγάλος αριθμός ετούντων άσυλο. Πρώτοι αυτοί μπορούν να αποδείξουν ότι δεν φίδονται αλτουρισμού και θέλουν να βοηθήσουν του ανθρώπου που έχουν ανάγκη στον τόπο του προτού αναγκαστούν να προσφύγουν στη δική μα βοήθεια. Στο ΙΑΚ γνωρίζουμε καλά το ΝΤΑΕΣ. Θα ετηθεί ολοκληρωτικά μόνο όταν η χώρα σταθεροποιηθεί και αναπτυχθεί και πάλι. Είναι εξόχω ευρωπαϊκό και προνοούμε να σταθεροποιούμε τα κράτη προτού να πρέπει να αντιμετωπίσουμε νέα μεγαλύτερα προβλήματα αύριο αναφορικά με το Ιράν. α υποστηρίξουμε ενεργά τις συμφωνίε μα. Α στηρίξουμε το κοινό συνεργατικό σχέδιο δράση. Ο, ο είναι μια όρημη δημοκρατία. Οι καταβάσει ελληνικέ διαδηλώσει αποτελούν δείγμα τη ποιότητα κοινωνία. Κατανοούμε ότι η κυβερνητική μετάβαση σε μια τεχνοκρατική κυβέρνηση θα επιτρέψει στη χώρα να κάνει τι απαραίτητε μεταρρυθμίσει και αναγνώριση εκλογέ. Η ευρωπαϊκή στάση προ τι χώρε τη περιοχή οφείλει να είναι η εσωτερική σταθεροποίηση με παράλληλη προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προσφορή του διεθνού δικαίου, η συνεργασία και το εμπόριο με ρήτρε αρισιμότητα. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Αρένα, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μακερίνη, 100%, 200% συμφωνώ με την δήλωση που κάνατε όσον αφορά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Όντως καίγεται εδώ και αρκετό καιρό και υπάρχουν ένα σωρό διεκδικήσεις που είναι λίγο πολύ ίδιες, κοινωνικές και για μια χρηστή διακυβέρνηση. Δεν ξέρω αν ήταν ο κύριος Γκετά ή κάποιος άλλος που το είπε. Όντως βλέπουμε δεξιά και αριστερά κυβερνήσεις οι οποίες ανταποκρίνονται με καταστολή στις διεκδικήσεις αυτές και πολύ συχνά με βία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ρόλο να παίξει με την εξωτερική της πολιτική για το σεβασμό του κράτους δικαίου και της πολυμερούς διάστασης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αντίθεση με την κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να συνεισφέρει στην αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή και να συνεχίσει να στηρίζει την ειρήνη και το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το είπαμε ότι η λύση στη Μέση Ανατολή θα περάσει από μη δημοκρατική μετάβαση που πρέπει να στηρίξουμε με το διάλογο όπως κάνετε εσείς, αλλά και με τη στήριξη και την προστασία των πληθυσμών εκεί. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κροσέλ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Η Μέση Ανατολή αρχίζει να διακρίνεται από διάφορες κρίσεις ε, που ρίχνουν ε, ε, σε ένα γκρεμό την περιοχή. Έχουμε την κρίση στο Ιράν, στο Λίβανο. Η λύση πολλών προβλημάτων βρίσκεται στα χέρια του Ιράν. Δυστυχώς πολλά κράτη στην περιοχή επηρεάζονται από την, περιοχή, από την πολιτική του Ιράν και από τους ήττες εκεί. Μετά από την αποτυχία της Ιρανικής Συμφωνίας, ε, το Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης ε, της περιοχής. Πρόκειται για μια βίαιη ρεαλπολιτικ που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κυρώσεις δεν αλλάζουν την κατάσταση δυστυχώς, ε, αλλά η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακυβεύεται. Οπότε απευθύνω έκκληση προς τον ε, νέο είπα το εκπρόσωπο να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την περιοχή ώστε να αποφευχθούν οι τεράστιες ροές μεταναστών. Ευχαριστούμε κύριε Σουρτασούν, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μογκερίνη. Έχουμε κοινωνικές διαμαρτυρίες στη Μέση Ανατολή τον τελευταίο καιρό. Λίβανος, Ιράκ, Ιράν μπορεί να μην φαίνεται αλλά έχουν πολλά κοινά. Λείπουν οι βασικές υπηρεσίες, υπάρχει διαφθορά και οι διαμαρτυρίες κατά των κυβερνήσεων στις τρεις αυτές ε, χώρες ε, οδήγησαν στην καταστολή δυστυχώς με αποτέλεσμα θανάτους ε, το ίντερνετ διεκόπη στο Ιράν και έτσι δεν μπόρεσε να ενημερωθεί ο κόσμος για το τι συμβαίνει. Χρησιμοποιείται η βία που οδήγησαν ακόμα και σε θανάτους διαδηλωτών που διαδήλωναν ειρηνικά. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην ελευθερία έκφρασης και στην ελευθερία ειρηνικής διαδήλωσης και να επιτραπεί η πρόσβαση στο ίντερνετ που απαγορεύτηκε στο Ιράν. Η αύξηση τώρα στην τιμή της βενζίνης στο Ιράν έχει επιπτώσεις ακόμα περισσότερο στην οικονομική κατάσταση, αλλά οφείλεται και στη στάση των Ηνωμένων που πιέζει ε, την Ιρανική οικονομία και ξέρουμε ότι θέτει και σε κίνδυνο την ε, πυρηνική συμφωνία. Οι κυρώσει, οι οικονομικές, οι άλλες, όπως είπα, οδηγούν στον υποφέρει ακόμα περισσότερο η καθημερινότητα των πολιτών εκεί δεν βάζει την κυβέρνηση του Ιράν μπροστά ε, στις ευθύνες του, κάτι το οποίο μας μας απασχολεί και ξέρω ότι σας απασχολεί και εσάς. Λοιπόν, πάντως από το Ιράν μέχρι το Λίβανο και μέσω του Ιράκ, οι ηγέτες των χωρών αυτών πρέπει να ακούνε τους λαούς και να βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής. Η ευημερία του κόσμου έχει πολύ μεγάλη σημασία και να σταματήσει η διαφθορά. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει να βοηθήσουμε στην προσέγγιση στην περιοχή, ώστε να συνοδεύσουμε και να λύσουμε ε, τα προβλήματα και κυρίως τις ρίζες που οδηγούν στην κατάσταση αυτή της χώρας για τις οποίες συζητάμε και οδηγούν και σε αστάθεια βέβαια στην περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Λίτση. Ενάμιση λεπτό. Πρόεδρε, κυρία Μογκερίνη, να πω ότι πέντε Ιταλοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν στο Κυρκούκ στο Ιράκ πρόσφατα ακριβώς λίγες μέρες πριν από την soprattutto nelle zone sciite. Si tratta di persone che chiedono lavoro e lottano contro la corruzione. Sono rimaste finora estranee alle Λίγες μέρες λοιπόν μετά από αυτό που είχε συμβεί στο παρελθόν στην Ασσύρια στο Ιράκ πολλαπλασιάζονται δυστυχώς ε, οι τρομοκρατικές απόπειρες. Το κράτος ε, το Ισλαμικό αναδιοργανώνεται. Δεν μπορούμε να μην, αντιδράσουμε. Ε, νομίζω ότι υπάρχει στην πλατεία του Ταχρήρ και ε, ίχνος του 1,5 σχεδόν των χριστιανών του Ιράκ, οι οποίοι κάποτε ήταν 1.300.000 και τώρα έχουν μείνει λίγοι εκατοντάδες χιλιάδες. Ακόμα και ο Τραμπ έχει χρηματοδοτήσει σωστά τις ε, χριστιανικές οργανώσεις. Ο ρόλος στο Ιράκ των ε, μειοψηφιών είναι πάρα πολύ ε, σημαντικός. Πρέπει να υποστηρίξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση την χριστιανική μειονότητα στο Ιράκ. Κύριος Βέμες, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόσωπε Μόγκερινη, αντί να κάνετε τεμενάδες στους μουλάδες και να αγωνίζεστε για να διαφυλάξετε τη συμφωνία με το Ιράν που απλά δίνει ε, προνόμια στο καθεστώς. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να υπερασπιστούν τον Ιρανικό λαό, να πετάξουν τη χιτζάμπ και να αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για ένα καθεστώς που ενδιαφέρεται περισσότερο για τους τρομοκράτες από ότι για το λαό του. Δεν, μπορούμε, δεν μπορεί να ανεχτεί τη διαφωνία, την ελεύθερη σκέψη ε, που δίνει διαταγή σε στρατιώτες να πυροβολούν κατά βούληση σε που καταστέλει εδώ και χρόνια και καταπιέζει του πολίτε του. Στι καρδιέ μα, εμεί οι Ευρωπαίοι, στεκόμαστε στο πλευρό των θαραλέων Ιρανών. Ε, χωρία Ισλάμι, ναι Μιχάη, ναι Μιχάη. Εμεί δεν θέλουμε Ισλαμική δημοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Βιλανούεβα Ρουίς, για ένα λεπτό παρακαλώ. Όχι μόνο βρίσκεται σε πολιτική τραχή η Λατινική Αμερική, αλλά και η Μέση Ανατολή και το Σουδάν και η Αλγερία, χώρες που περνάνε από σοβαρές κρίσεις. Πολλοί προσπαθούν να βάλουν χέρι στους τους και ο κόσμος ζητάει κοινωνική δικαιοσύνη εδώ και χρόνια. Ε, η απάντηση ήταν καταστολή και ακόμα μεγαλύτερο γεωπολιτικό χάος από την παράνομη παρέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράκ μέχρι την Ιγυρία και όλο και μην ξεχνάμε και την Παλαιστίνη, τη Δυτική Σαχάρα, τους Κούρδους. Κάθε μία από τις κρίσεις αυτές υποφέρανε μέχρι τώρα και εξαιτία τη εμπλοκή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση τι εγκαταλείπει αυτέ τι χώρε με καταστροφικέ συνέπειε. Η Ευρώπη θα πρέπει ανάμεσα στι στρατιωτικέ παρεμβάσει να φροντίσει να είναι μια δύναμη ανεξάρτητη σταθεροποίηση υπέρ τη δικαιοσύνη και υπέρ των ανθρώπων που διαδηλώνουν στον κόσμο και υπέρ τη ίδια ε, τη αποστολή και του μέλλοντο τη δικιά μα Υπήρου. Ευχαριστούμε κύριος Μπελαμή. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μογκερίνη, το είπατε. Η περιοχή αυτή για την οποία μιλάμε σήμερα, η Μέση Ανατολή, υποφέρει από μεγάλες εντάσεις και στην κατάσταση αυτή η Ευρώπη πρέπει να έχει τρεις στόχους. Πρώτον, να βοηθήσει τις χώρες αυτές που θέλουν τη δημοκρατία που θέλουν να πάνε σε ένα πιο ισχυρό κρατό δικαίου. Και σκέφτομαι εδώ όλου οι να πούμε και εγώ Γάλλο, του φίλου μα στο Λίβανο που πρέπει να υποφεληθούν από τη δικιά μα στήριξη στη μετάβασή του. Δεύτερο στόχο μα να διασφαλίσουμε τον ιστορικό μας ρόλο που είναι προστασία των μειονοτήτων. Και εδώ έχω υπόψη μου τις χριστιανικές μειονότητες. Εμείς πρέπει να τις προστατεύσουμε σε αυτή την περιοχή, αλλά και τους γεζιτή και όλους που κινδυνεύουν από τη βία και να φροντίσουμε να διασφαλίσουμε την ειρήνη και την προστασία όλων των ανθρώπων σε όποιο πιστεύουν. Και τέλος, ο τρίτος μας στόχος πρέπει να είναι να φροντίσουμε, όπως υπενθύμησε και ο συνάδελφος πριν από λίγο, οι εξελίξεις αυτές να μην ε, χειραγωγούνται από τον Ισλαμισμό που είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας σήμερα. Το ξέρουμε, ο τρόπος με τον οποίο το ριζοσπαστικό Ισλάμ θέλει να ελέγξει την περιοχή ε, επί τη ευκαιρία των ετοιμάτων για δημοκρατία πρέπει εμάς να μας καταστούν ιδιαίτερα προσεκτικούς. 13 ε, Γάλλοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στο Μαλί προχτές ακριβώς επειδή επολεμούσαν κατά του εχθρού αυτού. Και εσείς δείξατε στη Γαλλία τη στήριξή σας αυτή τη στιγμή υπέρθους, αλλά πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Οι χώρες μας δεν μπορούν από μόνες τους να βοηθήσουν, πρέπει ενωμένοι να έχουμε και στρατιωτικές δυνάμεις από κοινού για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Συγχρόνως πρέπει να έχουμε τα μέσα να δράσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, για παράδειγμα, ή μέσω μιας πιο μόνιμης δέσμευσης υπέρ της Ευρώπης. Τότε θα βοηθήσει την ειρήνη η Ευρώπη εφόσον φροντίσει να έχει αυτονομία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριος Μπενιφέη. μισή λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συζητάμε για χώρες εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους, οι οποίες όμως μοιράζονται αντίστοιχες μορφές διαμαρτυρίας από χιλιάδες κατοίκους που θέλουν καταπολέμηση της διαφθοράς και κοινωνική δικαιοσύνη. Ε, μοιάζει λίγο βέβαια με αυτά που συνέβησαν το 2011 και θυμίζω ότι παρά την αραβική άνοιξη δεν λύθηκαν τα διαφθορτικά προβλήματα. Ο Λίβανος υποδέχθηκε ε, σχεδόν το 30% του πληθυσμού του επιπλέον με τους Σύρους πρόσφυγες και έχει ένα κράτος το οποίο πρέπει να στηριχθεί ακόμα περισσότερο γιατί βρίσκεται στα όρια της καταστροφής οικονομικά. Είναι επίσης ε, και σημαντικός ο τρόπος ο οποίος ε, με τον οποίο μάλλον ε, ο στρατός της Συρίας χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες και επίσης άλλες καταστάσεις οι οποίες οδηγούν πολλές φορές στην απώλεια ανθρωπίνων ζώων και νομίζω ότι Θυμίζω εδώ και την επίθεση την οποία οργάνωσε τον ΤΑΕΣ και διεκδικεί τον ΤΑΕΣ εναντίον των Ιταλών στρατιωτικών, ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση των Αμερικανών και μετά από την προδοσία, το σκάνδαλο μάλλον που προκάλεσαν με την εγκατάλειψη των Κούρδων. Και γι' αυτό ευχαριστώ τη Μογκερίνη για τις προσπάθειες τις οποίες κάνει. Η κυρία Αλσαχλάνη να ξεκινήσω λέγοντας πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθήσαμε δύο φορές να περάσουμε ένα ψήφισμα για το Ιράκ και αποτύχαμε. Και θα ήθελα να ζητήσω από τα πολιτικά κόμματα γιατί μπλοκάρετε το ψήφισμα για το ε, ε, Ιράκ. Μιλάτε αλλά είστε όλο λόγια. Τώρα για την κυρία Μογκερίνη. Έχουμε μπροστά μας μια ιστορική επιλογή. Είτε θα στηρίξουμε τον λαό του Ιράκ ή θα στηρίξουμε την κυβέρνηση. Οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται. Ο λαός θα είναι πάντα εκεί όμως. Τι μέτρα συγκεκριμένα θα αναλάβετε για να βοηθήσετε τον πληθυσμό του Ιράκ να, να θέλουν να έχουν μια χώρα η οποία να ακούει αυτά τα οποία λένε, αυτό ζητάνε στις διαδηλώσεις του στην πλατεία Ταχρήρ. Να συγχαρώ εδώ τη θέση ε, του πρέσβη της Ένωσης στο Ιράκ για τις σωστές θέσεις τις οποίες παίρνει, επαναλαμβάνω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει αξιοπιστία στην περιοχή και η μόνη νομίζω που ε, μπορούμε να βοηθήσουμε, εξακολουθούμε ε, να βοηθήσουμε, είμαστε πάντα εμείς. Κύριος Τσίμνιο, 1,5 λεπτό. Αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ε, αναφέρω ένα επίγον πρόβλημα ασφαλείας που υπάρχει στην Ευρώπη και αποτελεί τεράστια ε, απειλή για την Ευρώπη. Οι μαχητές του Ισλαμικού κράτους που έρχονται από τη Σύρια και από άλλες χώρες, 4.000 ε, άνθρωποι έχουν ε, προσαρτηθεί στο Ισλαμικό κράτο στην Ευρώπη και δεν έχουμε αναπτύξει κάποια συγκεκριμένη στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε αυτού του τρομοκράτε. Θα έπρεπε να έχουμε τέτοια στρατηγική. Αυτή είναι μια πολιτική ε, Το, η κατάσταση στη Συρία κάνει το πρόβλημα πιο οξύ. Ε, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα ασφάλειας για το μέλλον τι θα κάνουμε με όλους αυτούς τους εγκληματίες ε, που βιάζουν, που σκοτώνουν με βιαιότητα, που δημιουργούν συμμορίες. Ε, τελικά είναι μικρές οι που επιβάλλονται από τα δικαστήρια στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα μοιραίο μήνυμα για τα θύματα αυτών των ε, ε, βιοπραγιών. Αυτοί οι τρομοκράτες πρέπει να τιμωρούνται αυστηρά. Δεν αξίζουν οποιαδήποτε λύπηση. Ε, θα πρέπει να οργανωθεί ένα ε, δικαστήριο εγκλημάτων πολέμου για τη Συρία. Οι τρομοκράτες είναι τρομοκράτες, είναι όλοι εχθροί μας. Θα πρέπει να λάβουμε τις ευθύνες μας. Μόνο έτσι θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τα θύματα. Όλοι εδώ θέλουμε ε, και έχουμε την ευθύνη για την ασφάλεια των πολιτών μας. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή την, να σταθούμε στο ύψος αυτής της ευθύνης. Ευχαριστώ η κυρία Κέμπα για ένα λεπτό. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επιτροπέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδίας για όλα όσα κάνατε. Σας ευχαριστούμε για τα πάντα, για τις προσπάθειές σας και για τη βοήθειά σας. Ευχαριστούμε για την βοήθεια προς όλους όσοι ε, ανεπλάξαν ε, σε αυτές τις υποθέσεις τους πολέμους στην αποσταθεροποίηση της περιοχής. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να έχει ένα πιο καλό ε, παγιωμένο σχέδιο δράση, όχι μόνο διπλωματικό αλλά και οικονομικό. Ένα σαφή δρόμο που να αφορά την Ιορδανία, το Λίβανο αλλά και το Ιράκ. Διότι αν πάτε να δείτε τι συμβαίνει στο Ιράκ, πολλές χώρες προσπαθούν να βοηθήσουν το Ιράκ. Οι Ούγγροι, για παράδειγμα, βοήθησαν στην ανοικοδόμηση ε, με 8 εκατομμύρια δολάρια και άλλα μέρη, τα Οπασίκα, Μπατέα, Μπατνάια. Αν ο κόσμος είχε που να επιστρέψει, θα επέστρεφε. Αυτή η αποσταθεροποίηση θα σταματούσε. Αυτό θα πρέπει να διασφαλίσουμε. Χρειάζονται συγκεκριμένα έργα τα οποία θα δείξουν ότι κάνουμε συγκεκριμένη δουλειά, ότι έχουμε απτές δράσεις. Είναι σημαντικό για την περιοχή. Ο κύριος Ρουίτ Ντεβέσε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε, τη εκπρόσωπε για το έργο σας και για την δήλωση που κάνατε σήμερα, την οποία στηρίζω. Αν ε, δούμε τι συμβαίνει στον ε, Ισλαμικό-Αραβικό κόσμο, την κατάσταση στην Αλγερία, στο Λίβανο, στο Ιράκ, στο Ιράν, θα μπαίναμε στον πειρασμό να σκεφτούμε ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας ε, δεύτερης αραβικής άνοιξης στο Λίβανο, στο Ιράκ, στο Ιράν, με τις διαμαρτυρίες, με αλλαγές στην κυβέρνηση στο Λίβανο και με καταστολή στην περίπτωση του Ιράν να παραδεχτεί. Νομίζω είναι σωστά αυτά που είπε και η συνάδελφο από το Ρινιού, ότι δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να τοποθετηθεί με ψήφισμα όσον αφορά το Ιράκ. Και ο επόμενο ύπατο εκπρόσωπο, ο κύριο Μπορέλ, θα πρέπει με μεγάλη σοβαρότητα να δει το ζήτημα των τριών αυτών χωρών για να καταλήξουμε σε κάποιες αποφάσεις όσο τις αφορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κιούτσουκ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σήμερα δεν έχουμε σταματήσει να ασχολούμαστε με την περιοχή όλο αυτό το καιρό που πλήττεται από συγκρούσεις, πολέμους κλπ χωρίς να βλέπουμε να αλλάζει τίποτα για τον κόσμο που ζει εκεί. Αντίθετα, όλο και περισσότερη τρομοκρατία με πάρα πολλά θύματα. Έπειτα, ε, διαδηλώσεις που καταλήγουν σε νεκρούς. Οι πολιτικοί εκεί δεν θέλουν να δεχτούν ε, την πραγματικότητα και να δώσουν ελπίδα ε, στον κόσμο. Είναι μια θλιβερή πραγματικότητα. Μια εφημερίδα του Ιράκ έθεσε το εξή ερώτημα κατά σύμπτωση. Αν μας σκοτώσετε όλους, τότε ποιον θα έχετε πάνω στον οποίο να κυριαρχήσετε. Έτσι λοιπόν ζητάμε από τις αρχές των χωρών αυτών να σταματήσουν τη βία σε βάρος των διαδηλωτών αμέσως και να ανοίξουν ε, τις ε, πόρτες. Οι βουλευτές ε, θα πρέπει να εκπροσωπούν το δημόσιο συμφέρον και να αλλάξει ο τρόπος που ασκούν την πολιτική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάννη, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να ακούσουμε τον θυμό των Λιβανέζων. Αλλά θα πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί, γιατί όλες οι εξελίξεις στο Λίβανο έχουν να κάνουν και με τις διαφορετικές θρησκευτικέ κοινότητες και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι χριστιανοί οι οποίοι απειλούνται όλο ιδιαίτερο στην περιοχή. Έτσι λοιπόν, ω Ευρωπαίοι εκλεγμένοι, θα πρέπει να ρωτηθούμε τι γίνεται με τα εκατομμύρια τα οποία φτάνουν στο Λίβανο για βοήθεια σε αυτή τη χώρα. Να, η επιστολή ενό εκλεγμένου ερετού από την Τρίπολη του Λιβάνου που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει έναν σταθμό επεξεργασίας αποβλήτων που δεν λειτουργήσε ποτέ. Γιατί οι δωρητές δεν ελέγχουν τι γίνεται, γιατί τα χρήματα αυτά δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους και γιατί η Ευρώπη δεν κάνει τίποτα για να ελέγξει την κατάσταση και να φροντίσει να μην υπάρχει διαφθορά. Να λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε προ όφελο των Λιβανέζων. Τα χρήματα τα οποία δίνουν οι Ευρωπαίοι για να του βοηθούν να πηγαίνουν πραγματικά στον κόσμο και όχι να χάνονται στη διαφθορά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζαχράντιλ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην προηγούμενη συζήτηση είπα ότι το Ισραήλ είναι ο βασικός στρατηγικός μας εταίρος από την ε, περιοχή. Αλλά το Ιράν είναι ο στρατηγικός μας αντίπαλος στην περιοχή. Και αυτό που διαπιστώσαμε για χρόνια ολόκληρα είναι η απόπειρα του Ιράν να επιβάλλει την ηγεμονία του στην περιοχή. Είδαμε τι έγινε με το Ιράκ. Επίσης, ε, ε, η παρουσία και η επέμβαση της Συρίας στο Λίβανο υπονομεύοντας την εσωτερική συνοχή της περιοχής. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πολιτική του Ιράν. Θα πρέπει να στηρίξουμε την αντιπολίτευση και να, να είμαστε αποφασισμένοι στη θέση μας και ε, για να προσπίσουμε τα συμφέροντά μας στην περιοχή. Θα πρέπει να κάμψουμε το Ιράν. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχισμένης στρατηγικής μας στην περιοχή. Η κυρία Γκούτελαντ, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Μογκερίνη, ακούμε σήμερα δηλώσεις διεθνών οργανισμών που λένε ότι το Ιρανικό κράτος ε, ε, αντιμετωπίζει βία τους διαδηλωτές. Πολλοί σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν και συνελήφθησαν. Άνθρωποι οι οποίοι διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους. Απαράδεκτο να σκοτώνονται, να τραυματίζονται, να συλλαμβάνονται, να αντιμετωπίζονται με τέτοια κτηνοδία. Και κόβουν και το ίντερνετ. Ε, μιλάμε δηλαδή για παραβιάσεις ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. και ταυτόχρονα γράφουν ε, Twitter από εδώ και από εκεί και λένε ότι δεν υπάρχει πρόσβαση σε διάφορα βασικά αγαθά. Εγώ και οι συναδελφοί μου καταδικάζουμε τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν και αναμένουμε σοβαρή αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνατε κυρία Μογκερίνη και ελπίζω γρήγορα να γίνει κάτι σε σχέση με το Ιράν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χόλβορ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ σαν αντιπρόεδρο ε, τη αντιπροσωπεία με το Ιράν. Θα ήθελα να επικοινωνήσω σε αυτή τη χώρα και μιλάω ω υποστηρικτή ε, του σχεδίου δράση ε, του κοινού. Είμαι κατά των κυρώσεων των Αμερικανών που δεν, δεν πρέπει να υπονομεύουν τους μετριοπαθείς είναι όμω όλο και πιο γρήγορα, δύσκολα τα πράγματα κάθε φορά που το Ιράν παραβιάζει του ε, διεθνεί κανόνε. Ε, η βία ήταν εντελώ ε, δυσανάλογη με την οποία, την οποία αντιμετωπίστηκαν οι διαδηλωτέ. Έχουμε περίπου 100 νεκρού, χίλιου συλληφθέντε. Ε, χαίρομαι που θα υπάρξει μια νέα κοινή επιτροπή, όμω πρέπει πραγματικά να καταδικάζουμε Αυτέ τις φρικαλαιότητε όποτε και όπου συμβαίνουν. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μογκερίνη για την ε, ε, ε εντυπωσιακή της παρουσία εκεί και ε, εδώ και για την ε, υπομονή της βέβαια ελπίζω το ίδιο να μπορέσει να κάνει και ο, ο, ο επόμενος ε, ο διάδοχός σας και ελπίζω να μην είμαστε ξένη χώρα εμείς στον Βασίλειο τότε Βίες ε, διαδηλώσεις έχουν συνταράξει το Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τίποτα. Έχουμε μία ύπατη εκπρόσωπο. Τι κάνατε κυρία Μογκερίνη, τίποτα. Η Ευρώπη έχει επιτρέψει τα τελευταία χρόνια τα ανεπίτρεπτα ε, εκτελέσεις, ε, βασανιστήρια και όλα αυτά και τρομοκρατία στο Ιράν. Μεταξύ δε των καταδικασμένων υπάρχουν 90 γυναίκες. Και πού είναι λοιπόν οι φεμινίστριες εδώ πέρα του μύτου, αντί η Ευρώπη να μιλάει για τον ε, εξυγχρονισμό και την ελευθερία, αποφάσισε να σιωπήσει λόγω του πετρελαίου. Λοιπόν, έχουμε απλά πράγματα, νεκρούς, ε, τραυματίες ε, και λογοκρισία στο ίντερνετ. Γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν πλέον Ισλαμική Δημοκρατία. Πότε η Ευρώπη επιτέλου θα υπερασπιστεί την ελευθερία και τη δημοκρατία. Λόπε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, να ευχαριστήσω και την είπατε εκπρόσωπο. Είμαστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα για τι ε, πολύ σημαντικέ διαδηλώσει που έλαβαν χώρα σε διαφορετικού λόγου σε διάφορε περιοχέ. Στο Λίβανο, στο Ιράκ, στο Ιράν. Να εξηγήσουμε όμω κάποια κοινά σημεία ε, σε αυτές τις εκδηλώσεις. Υπάρχει τεράστια δυσαρέσκεια, κοινωνική δυσαρέσκεια, δεν υπάρχουν ευκαιρίες, δεν υπάρχει πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, θέλουμε, θέλουν μια οικονομική ανάπτυξη να φτάνει σε όλο τον πληθυσμό. Υπάρχουν βεβαίως και σειράξεις που τα τελευταία χρόνια δυστυχώς ε, έχουν ε, πλήξει του τοπικού πληθυσμού, υπάρχει μια πόλωση σε περιφερειακό επίπεδο. Ε, οι θεσμοί εκεί δεν είναι αρκετά συμπεριληπτικοί. αυτό που ζητούμε και αυτό που προσπάθησε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια είναι πρώτον να υποστηρίξουμε αυτά που κάνει η διεθνής ε, ε κοινότητα για να βελτιωθεί η κατάσταση, όπως συμφωνία για τα, για πυρηνικά. Να ζητήσουμε από το Ιράν να λογοδοτήσουν αυτού του αυτούς τους οι με νεκρούς. Και επίσης να υποστηρίξουμε μια χώρα όπως ο Λίβανος που υποδέχεται πάρα πολλού πρόσφυγες και έχει πολύ σημαντικά οικονομικά προβλήματα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Μαρία Ροντρίγκε ράμο. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώ η ομιλήτρια. Παρακαλώ ανάψτε το μικρόφωνο σας γιατί δεν ακούγεστε. Συγγνώμη, ξαναρχίζω. Έλεγα λοιπόν, κυρία Μογκερίνη, ότι σας ευχαριστώ θερμά για το έργο σας και για τις προσπάθειες και την προσήλωση που δείξατε όλα αυτά τα χρόνια. Οι διαμαρτυρίε ε, που γίνονται στην περιοχή ε, είναι διαμαρτυρίε όπου ο κόσμος ζητά περισσότερη δημοκρατία, ελευθερία, κοινωνικά δικαιώματα και αυτές οι αναταραχές ε, καταστάλησαν με μεγάλη βαναυσότητα με τη χρήση πυροβόλων όπλων εις βάρος του άμαχου πληθυσμού, εις βάρος των άοπλων πολιτών. Και μας είπαν ότι έχουμε δεκάδες για να μην πω εκατοντάδες νεκρούς. Βάσει της Δεθνούς Αμνηστίας έχουμε 4.000 τραυματίες, 10.000 κρατούμενους, λιθέντες. Παρόλο που η α, χώρα επέβαλε ένα εμπάργο στις πληροφορίες και έκλεισε το διαδίκτυο. Επίσης είναι τεράστια επίση προς τις γυναίκες ε, τις ε, στελιτεύουν ως υπεύθυνε υπέτειες και υποκινήτριες των ε, αναταραχών αυτών. Ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Διεθνή Κοινότητα να καταδικάσει, να καταγγείλει και να στυλιτεύσει αυτά τα περιστατικά, να ζητήσει από τι Ιρανικέ Αρχέ να σταματήσουν την καταπίεση και την καταστολή και να απευθύνουμε έκκληση προ ένα γνήσιο πολιτικό και δημοκρατικό διάλογο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριο Λάρ Μπέρκ. Για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, είπατε εκπρόσωπε, θα περιοριστώ στην κατάσταση στο Λίβανο. Όλοι είδαμε πώς διαμορφώθηκε η κρίση με την παρέτηση της κυβέρνησης του Λιβάνου λόγω των διαδηλώσεων και με την αδυναμία σχηματισμού νέας κυβέρνησης. Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται η Χεσμολά μια τρομοκρατική οργάνωση και πίσω από την Χεσμολά είναι ο χρηματοδότης της η Ιρανική κυβέρνηση. Ο Λίβανος υποφέρει λόγω των ξένων παρεμβάσεων και τη σύγκρουση συμφερόντων στο έδαφος του. Η Χεσμολά είναι εκπρόσωπος του Ιράν και αποσταθεροποιεί τη χώρα που ούτως ή άλλως δεν είχε και πολύ μεγάλη σταθερότητα η Χεσμολά και το κίνημα Αμάλ επιτίθενται σε διαδηλωτές ε, στην Βηρητό και προσπαθούν να διατηρήσουν την επιρροή του Ιράν. Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν θα δεχτεί άλλες επιθέσεις ε, της Χεσμολά στην επικράτειά του. Πρέπει λοιπόν ε, να μην επιτρέψουμε ο Λίβανος να ξαναγίνει πεδίο μάχης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος ε, Ανδρέας Σίντερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε, κυρία Ήπατη Εκπρόσωπε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερος για τις πολλές ε, πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει και την δουλειά που έχετε κάνει και την επίσκεψή σας βεβαίως για να επιτύχετε μια συμφωνία με το Ιράν. Αλλά βλέπουμε συγκλονιστικές εικόνες τελευταίες μέρες ε, από το Ιράν. Ταραχές, διαδηλώσεις και η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη για τον λαό. Έχουμε εκατοντάδες ε, νεκρούς, ε, χιλιάδες ε, συλληφθέντες. Η Ιρανική κυβέρνηση πρέπει να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία λόγου, την ελευθερία του συνέρχεστε, την ελευθερία να διαδηλώνει ο κόσμος και βεβαίως το ελεύθερο διαδίκτυο. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν αποκλιμάκωση και να επανέλθουν και οι δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η κρίση θα πρέπει να αποκλιμακωθεί και να μην ρίχνουμε άλλο λάδι φωτιά όπως κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Έλενα Γιόντσεβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μου για την κλιμακόμενη